ή μπορούμε να θρέψουμε τους συμπολίτες μας ή τότε δεν έχει νόημα να υπάρχει Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μποβέ. Η ψηφοφορία της έκθεσής σας θα λάβει χώρα στις 12, σε λίγα λεπτά δηλαδή. Και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της μερισιάς διάταξης που είναι η έκθεση του κυρίου Πάτρι Τσέλο για τη διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισηγήτης έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Το διάστημα είναι στην επικαιρότητα. Ιδιαίτερα μετά από τους δύο δορυφόρους για το Γαλιλαίο που ανέλαβαν υπηρεσία μετά την εκτόξευσή τους από τη βάση του Κουρού. Είναι ένα πρώτο βήμα για την επίτευξη της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην δορυφορική πλοήγηση. Νομίζω ότι είναι μια όθηση που δόθηκε από το άρθρο 199 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο ξεκαθαρίζει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και την εγκαθίδρυση όλων των πολιτικών των εθνικών στον τομέα του διαστήματος έτσι ώστε να ευνοηθεί η επιστημονικοτεχνική πρόοδος και η ανταγωνιστικότητα η βιομηχανική. Ο στόχος ο οποίος ορίζεται από τη συνθήκη αναγνωρίζει τη σημασία που έχει το διάστημα και στον τομέα των υπηρεσιών και στον τομέα των οικονομικό και τον στρατηγικό και θα πρέπει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι λειτουργική για να μπορέσει να ανταγωνιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τους διεθνείς ανταγωνιστές της. Νομίζω ότι η βάση μας δίδει την κατάλληλη βάση για να πετύχουμε τους στόχους μέσω από τους οποίους η εθνική, η οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες για την εφαρμογή των πολιτικών τις οποίες θα αποφασίσουμε. Και στα πλαίσια της ΙΤΡΕ προχωρήσαμε στην διαμόρφωση της πρότασης για την διαστημική πολιτική της Ένωσης προς όφελος των πολιτών. Ελπίζω η τελική διατύπωση του κειμένου να σέβεται τις φιλόδοξες προτάσεις τις οποίες θελήσαμε να συμπεριλάβουμε. Αναφέρομαι κυρίως στην διαφορετική αντιμετώπιση δύο στρατηγικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής, το Γαλιλαίο και το Τζέμες. Νομίζω ότι η εμπιστοσύνη την οποία έχει δείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Γαλιλαίο είναι απόλυτα δικαιολογημένη και υπό το φως των επενδύσεων που έχουν διατεθεί μέχρι τώρα άνω των 3,5 δις και λόγω του στρατηγικού χαρακτήρα και το GMS απαιτεί ισότιμη αντιμετώπιση και ε, οικονομική και πολιτική. Μόνο αξιοποιώντας πλήρως τέτοιου είδους προγράμματα μπορούμε να εγγυηθούμε την τεχνολογική ανεξαρτησία και την πολιτική στη συνέχεια ανεξαρτησία της υπήρους μας, ωφελώντας κοινωνικά και οικονομικά τους πολίτες μας. Γι' αυτό λοιπόν η έκθεση της Επιτροπής Ήτρε που θα ψηφιστεί σύντομα ε, είναι θετικό, αλλά λυπάμαι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αποφάσισε να μην χρηματοδοτήσει το GMS στα πλαίσια του πολιετούς χρηματοδοτικού προγράμματος 2014-2020 γιατί η έλλειψη ενός τέτοιου προγράμματος επενδύσεων θα καταστήσει άχρηστες τις επενδύσεις που μέχρι τώρα έχουμε κάνει. Είναι σαφές λοιπόν ότι η στρατηγική την οποία θα προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαχειριστικές πλευρές των προγραμμάτων Galileo και GMS είναι απαραίτητο να οργανώσουν με σωστό τρόπο την διαχείριση αυτή και να περιορίσουν το κόστος. Στα πλαίσια της έκθεσης υπογραμμίζουμε την ανάγκη που υπάρχει η Ευρώπη να πρικιστεί με την δική της μορφή παρέμβαση στην διαστημική της διάσταση και οι εμπορικές σχέσεις με τις τρίτες χώρες να εδράζονται σε μια σχέση πλήρους αμοιβαιότητας αποτρέποντας καταστάσεις μονοπωλιακές και προμήθειας υπηρεσιών από έξω ευρωπαϊκούς ε, παράγοντες ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι εκτοξευθές ε, δορυφόρων. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε και την ερευνητική δραστηριότητα ενός φιλόδοξου προγράμματος το οποίο ελπίζουμε να δώσει τις απαντήσεις τις οποίες φιλοδοξεί να έχει ο Ευρωπαίος πολίτης. Πρέπει να βλέπουμε μακριά στην διαστημική πολιτική και να μην αγνοούμε τις ανάγκες της βιομηχανίας. Στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης είναι απαραίτητο η Ένωση να στηρίξει οικονομικά το παραγωγικό κομμάτι της διαστημικής βιομηχανίας διατηρώντας άτρωτη την ανταγωνιστικότητα της υπήρου σε ένα παγκόσμιο σύστημα ολοένα πιο ανταγωνιστικό. Μόνο εάν προσφέρουμε στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία απτές προοπτικές ανάπτυξης, τότε μόνο και αυτή θα επενδύσει σε ανθρώπινους πόρους και σε τεχνολογίες μακροπρόθεσμα. Μόνο η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία θα διατηρήσει την ηγετική της θέση και μόνο τότε η Ήπειρός μας θα παραμείνει πρωταγωνιστής σε αυτόν τον νευραλγικό τομέα. Προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν σαν εισηγητής για την Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική συνεχίζω την προσπάθειά μου θεωρώντας ότι μια θετική ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμβατή με το άρθρο 199 της νέας συνθήκης θα δώσει εγγυήσει για την τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη και την αηφόρο ανάπτυξη της συγκεκριμένης πολιτικής, μιας πολιτικής απαραίτητης για την Ένωση. Ευχαριστώ συνάδελφε Πατριτσέλο. Διαδικασία Catch the Eye. Πρώτος ομιλητής. Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. Sazada. Αγαπητοί συνάδελφοι, ορισμένες φορές δεν αντιλαμβανόμαστε το ότι και τα διαστημικά προϊόντα και οι δραστηριότητε που έχουν να κάνουν το διάστημα είναι σημαντικοί παράγοντε ανάπτυξης για τις κοινωνίες μα. Και για μένα η διαστημική τεχνολογία θα έχει ως μεγαλύτερο όφελο την τεχνολογία των ενέργων μεταφορών. Η ευρωπαϊκή εθέρεση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. και είναι πολύ σημαντικό να ρυθμιστεί η εναέρια κυκλοφορία έτσι περαιτέρω. Οι νέες τεχνολογίες θα φέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια για προστασία στις ε, αεροπορικές μεταφορές. Τα οικοσυστήματα δε και η ανείχνευση αντικειμένου σε πραγματικό χρόνο είναι κάτι πολύ θα γίνει πραγματικότητα. Το Θα ήθελα να γίνονται περισσότερε συνεδριάσει για το θέμα το διαστημικό και το Συμβούλιο δεν έχει εκφραστεί πολύ συχνά. Θα ήθελα να συζητιέται το θέμα πολύ ε, πιο συχνά. Κύριε Φατικά. Πρόσβαση στις ε, υποδομές. Πρέπει να υπάρχει επιτάχυνση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και ιδίως με ΙΠΑ. Η Ιαπωνία, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Χιλή, Αργεντινή και Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Πρέπει να στηρίξουμε την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της συστημικής πολιτικής να εξασφαλίσουμε τη τεχνολογική πρόοδο, τη βιομηχανική ε, πρόοδο, την ανταγωνιστικότητα για να δημιουργηθούν νέε θέσει εργασία στην Ευρώπη. Θα ζητήσουμε από την Κομισιόν να στηρίξει και τι μικρομεσαίες επιχειρήσει ώστε να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την καινοτομία στον τομέα του GNSS και, στο, και στην καινοτομία. Και το έγκνος θα πρέπει να καλύπτει όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Θέλουμε να νοποιήσουμε ε, τον εναέριο χώρο. Και βέβαια και αυτά να εφαρμοστούν και στην Ανατολική Ευρώπη. Παρακαλώ να είστε πιο αργοί όταν λαμβάνετε το λόγο, γιατί δεν μπορεί να σα παρακολουθήσουν οι διερμηνεί. Συνάδελφο Πάσκα είναι επόμενος ομιλητή. Vážený pán Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, ε, κυρίως εστιάζουμε στο GMES για την παρατήρηση της γης και το πρόγραμμα Galileo. Τι περιμένουμε από το Galileo στο άμεσο μέλλον να παρέχει υπηρεσίες ε, προς το ευρωπαϊκό κοινό. Από το 2014 και μετά θα ξεκινήσουν δοκιμές ε, για να δούμε κατά πόσον έχει σκοπιμότητα να υπάρχει αυτό το σύστημα και κατά πόσο είναι διαλειτουργικό με το GPS και άλλα συστήματα τα οποία ήδη ισχύουν θα μπορούμε να συμμετέχουμε και στη διεθνή συνεργασία των διεθνών συστημάτων δορυφορικής απλοήγησης. Τον Καλλιλέο μπορεί να παράσχει ωφέλη σε σχέση με ανταγωνιστικά συστήματα. Έτσι θα έχουμε και τα ε, απαραίτητα οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη από αυτό. Αλλά στρέφουμε προς την Κομισιόν με το εξή ερώτημα. Πώς πρέπει να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα παρατήρησης της γης GMES από το 2014 και μετά. Διακόπτε το μιλητής. Ο κύριος Μπρόνς τώρα έχει το λόγο. Thank you. Political states. Σας ευχαριστώ. Πολιτικά κράτη που θέλουν κάτι να, να παρουσιάσουν ε, θέματα πολύ σημαντικά. Παραδείγματο χάρη είναι ε, τον, η Ισπανία που ενώθηκε υπό τους χριστιανικούς ε, βασιλείς και ο, ο Χριστόφορος ξεκίνησε μετά ε, για να κρύψει πράγματα που δεν ξέραμε ότι δεν γνωρίζαμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να κάνει κάτι παρόν. Νέα προϊόντα, νέες ε, γνώσεις και ε, χρήματα για, την, ε, για το διάστημα. Η πραγματική κοινωνία είναι να δοθεί σε μια πολιτική μονάδα έτσι κάποια αξία. Προσπαθεί δηλαδή με τη διαστημική πολιτική να εδραιώσει θέση τη στο διεθνή σκηνή και να αποδείξει την ανεξαρτησία της. Ανεξαρτησία της Ένωσης σημαίνει δική μας σκλαβιά. Ευχαριστώ κύριο Πέτρο Λούχαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην Υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ συζητάμε ε, πολλές φορές την διαστημική στρατηγική, ιδίως σε ό,τι αφορά ε, την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή της διαστημικής στρατηγικής για να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο διεθνές προσκήνιο. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η βιομηχανική συνεργασία στη διαστημική πολιτική με τρίτε χώρε. Χρειαζόμαστε τη ΣΥΠΑ, χρειαζόμαστε την Ιαπωνία, την Κίνα, την Ινδία και άλλε χώρε οι οποίε έχουν πολύ μεγάλη δύναμη στον τομέα αυτό. Θα πρέπει επίση να προσελκύσουμε περισσότερο ιδιωτικό κεφάλαιο, κεφάλαιο από τον ιδιωτικό τομέα για το πρόγραμμα GMS e της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε επιτύχει. Τέλος, αλλά και εξίσου σημαντικό είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις επενδύσεις για να ε, ολοκληρωθεί το σύστημα Γαλιλαίο. Θα ήταν λάθος να χαθεί η όθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Ευχαριστώ. Βιτόριο Πρόντι. <coughs> Ευχαριστώ Επίτροπε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλάμε για πραγματικές ευρωπαϊκές υποδομές, απαραίτητες για την ολοκλήρωση και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών, ιδιαίτερα το GMS, είναι απαραίτητο για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και για τον έλεγχο των συνεπειών της υπερθέρμανσης του κλίματος και για τη βελτίωση ακραίων, ε, ε, διάγνωσης ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων πρέπει να συμπεριληφθεί στο πολιετές χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, τότε θα πρέπει να εισάγουμε στην περίπτωσή τους τα project bonds, τα ομόλογα που έχουν αντισυγκυριακή θα έλεγα σημασία, γιατί αυτά είναι η πραγματική επένδυση στο μέλλον και την, την επένδυση αυτή θα την αποσβέσουμε τάχιστα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Βιτόριο. Ήταν ο τελευταίο ομιλητή ο κύριο Πρόντι. Για να κλείσει τη συζήτηση, λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριο Ταζιάννη, ο επίτροπο. Θεωρώ ότι η διαστημική πολιτική είναι πολύ σημαντική για μένα τον ίδιο σαν επίτροπο. Οι υπηρεσίες αυτές ήδη παρέχουν στου πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωση υπηρεσίες Θεωρώ επίσης ότι ο βιομηχανικός τομέας, ο τομέας της βιομηχανίας, γιατί θυμίζω ότι υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις που ασχολούνται με το θέμα αυτό, ένα θέμα που άπτεται αυτού που ονομάζουμε η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να αναπτυχθεί με σωστό τρόπο επί τη βάση της εσωτερικής της αγοράς και με πραγματικές οικονομικές βάσεις. Συνεπώς λοιπόν ευχαριστώ τον κύριο Πατριτσέλο για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Ευχαριστώ και το Κοινοβούλιο και τα μέλη του Κοινοβουλίου όπως τον κύριο Πρόντι για την υποστήριξη των μέτρων που παίρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνούμε πλήρως όταν ζητάμε να υπάρξει μια διαστημική πολιτική πράγματι ανταγωνιστική ε, για την πολιτική μας. Τα αποτελέσματα τα οποία πετύχαμε τους τελευταίους μήνες είναι θετικά. Το έγνος έχει αρχίσει να λειτουργεί. Τον Οκτώβριο εκτοξεύσαμε από το Κουρού την Γαλλική Γουλιάνα τους δύο πρώτους δορυφόρους για την εφαρμογή του προγράμματος Γκαλιλαίο. Την ίδια μέρα της εκτόξευσης ξεκίνησα και την διαδικασία εγώ για την απόκτηση οκτώ νέων δωροφόρων και την 1η Φεβρουαρίου θα ανακοινώσω τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την προμήθεια και άλλων περαιτέρω δορυφόρων για το σύστημα Γαλιλαίος. Ο χρονισμός αυτός σε σχέση με τις προβλέψεις για την εξέλιξη του συστήματος μας επιτρέπει να εξοικονομούμε περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις του 2011 από την διοργανική ομάδα ε, δηλώσεις που είχαν κατατεθεί και στο Κοινοβούλιο στα πλαίσια της ανακοίνωσης που είχαμε κάνει για τη διαστημική πολιτική. Το Γκαλιλαίο όμως προχωρά. Πρόθεσή μου είναι οι υπηρεσίες που παρέχει το Γκαλιλαίο να είναι πλήρως λειτουργικές το τέλος του 2014 και το πλήρες σύστημα με 30 δορυφόρους να λειτουργεί μέχρι το τέλος του 2020. Λοιπόν, για την εφαρμογή του προγράμματος Γαλιλαίο και στα πλαίσια των προοπτικών των οικονομικών που παρουσιάσαμε προς το Συμβούλιο προβλέπουμε επενδύσεις περίπου 7 δις ευρώ. Αυτά προβλέπονται περιλαμβάνοντας και το 1,5 δις για την εκτόξευση των δορυφόρων και τα υπόλοιπα για την τεχνική διαχείριση και την παραγωγή των υπηρεσιών. Αυτή τη στιγμή λειτουργήσει τον Γαλιλαίο, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε έσοδα που μπορεί να φτάσουν και τα 90 δις. Τώρα σχετικά με αυτά που είπε ο Πατριτσέλο για το GMS η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια ανακοίνωση, νομίζουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, όμως προτείναμε να δημιουργήσουμε ένα μέσο χρηματοδότησης ad hoc εκτός κοινοτικού προϋπολογισμού, στα πλαίσια της Ένωσης βέβαια, μετά από μια συμφωνία των 27 κρατών μελών. Αντιμετώπισα το θέμα αυτό και στα πλαίσια της τελευταίας συνεδρίασης του Συμβουλίου για το διάστημα. Αναφέρθηκα επίσης το θέμα και στα πλαίσια του Συμβουλίου για την ανταγωνιστικότητα. Γιατί κάναμε την πρόταση αυτή. Κοιτάξτε, γνωρίζουμε ποια είναι η δημοσιονομική κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαν να είχαν πιο ανταγωνιστικές, θα έλεγα, επιλογές αλλά παρόλα αυτά η απάντηση δεν είναι αυτή την οποία όλοι ελπίζαμε. Έχουμε καταλήξει λοιπόν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε εμείς να χρηματοδοτήσουμε μέσω του προϋπολογισμού όλες τις δράσεις τις οποίες προβλέπουμε για τα επόμενα έτη και γι' αυτό ακριβώς και πέραν της πεποίθησης την οποία έχουμε Ε, για το ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί σωστά η διαστημική πολιτική και να χρηματοδοτηθεί σωστά το GMS το οποίο πράγματι θα βοηθήσει και τη διασύνδεσή μας και με άλλες χώρες στον υπόλοιπο κόσμο. Ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας συνεργαστήκαμε στους τομείς αυτούς και με την Αφρικανική Ένωση και με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, ως έχουν τα πράγματα, τα προβλήματα παραμένουν δημοσιονομικά και εξ αυτού και η δική μας επιλογή. Λοιπόν, η διαστημική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των, των οικονομικών προοπτικών και τον, του μεγάλου πακέτου των 80 δις ευρώ που προορίζονται για την έρευνα και την καινοτομία. Αποφασίσαμε αρκετά από τα χρήματα αυτά να τα επενδύσουμε στον τομέα του διαστήματος. Πρόκειται δηλαδή για μια επιπλέον ε, προστιθέμενη αξία την οποία θέλουμε, ε, με την οποία θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες της διαστημικής πολιτικής έτσι θα καλύψουμε τους στόχους τους οποίους θέτει και η έκθεση Πατριτσέλο. Νομίζω ότι η συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει σημαντικό και όλοι νομίζω ότι έχουμε κοινούς στόχους σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ λοιπόν. Κλείνουμε την συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει από τις 12 και μετά, σε λίγα λεπτά. Το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είναι η έκθεση για το πώς θα αποφύγουμε τη δαπάνη, τη σπατάλη των τροφή.